Υπάρχουν ε, ένα ψήφισμα από πέντε ομάδες του κ. Κομπένικ, Άλμπερτ και Πίτι Χόφερ. με τον... Ε, Περνάμε την ε, τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, ψηφ... κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι τι ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13 προς 36. Με 11 αποχές. Μετά έχουμε τροπολογία 1. Ονομαστική κλίση Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 8 υπέρ 45 κατά. 9 αποχές. Περνάμε τώρα στο σημείο 4, το αρχικό κείμενο, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά η φιλή σκέψη α, τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 14 ψήφοι υπέρ, 32 ψήφοι κατά. Απορρίφθη. 17 αποχέ υπήρχαν. Περνάμε στην απολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ετρολογική σκέψη ε. Τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 8 ψήφοι υπέρ, 40 κατά. Υπήρχαν και 16 εποχέ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σύνολο τη πρώτη ψηφίσματο. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές με λίγες ψήφους κατά και λίγες αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία 6 προτάσεων ψηφίσματος για το Μεξικό. Υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα από 5 πολιτικές ομάδες. Παράγραφος 1, τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ο φοφορίας. Απορρίπτεται. 8 ψήφοι υπέρ, 54 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τι ψηφοφορίε. Απορρίπτεται. 7 ψήφοι υπέρ, 54 κατά. Μία αποχή υπήρχε. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 8. Ποιο μπορεί να συμφωνήσει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παραγραφή 11, καταρπολογία 4, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 7 ψήφοι υπέρ, 54 κατά. Μία αποχή. Στην παραγραφή 12, τροπολογία 5, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι, πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται 6 ψήφοι υπέρ, 54 κατά 2 απόχέ. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 7 ψήφοι υπέρ, 55 κατά και μία αποχή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Στο σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. 57 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 3 αποχέ. Εγκρίνεται το ψήφισμα αυτό. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. 5 προτάσει ψηφίσματο για την Νότιο Κορέα. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία. Μπορούμε να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 50 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 4 αποχέ. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Έλαβα στην πρώτη ανάγνωση ε, και, πέντε, και την τοποθέτηση των ζώων από αυτών σε πέντε κείμενα. Θα βρείτε στα πρακτικά του τίτλους η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου αρχίζει αύριο, 12 Μαρτίου 2010. Τα πρακτικά τη τρέχουνα συνεδρία θα υποβληθεί στην αρχή τη επόμενη συνεδρία Συνόδου στο Κοινοβούλιο και αν δεν υπάρχει καμία διαφωνία θα ε, θεωρήσω τα ψηφίσματα που εγκρίναμε σήμερα θα προωθηθούν στους ενδιαφερόμενους. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανένας. Διακόπτεται εδώ η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή και σίγουρη επάνω επάνωδο. Oh,